Witam Państwa na popołudniowej sesji. Καλώ ήλθατε, συνάδελφοι. Καλώ ήλθατε στην απογευματινή μα συνεδρίαση. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Ας ξεκινήσουμε τις ε, απογευματινές μας εργασίες με τις ψηφοφορίες. Έχουμε την πρώτη έκθεση για την ε, προστασία και φροντίδα των εκτρεφόμενων κουνελιών. Ε, Στέφαν Εκ, έχουμε 30 συμβασμούς. Κύριε Εκ, έχετε το λόγο για να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη συνάδελφοι. Θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές, ε, τα γραφεία τους, τους συμβούλους τους ε, για την πολύ καλή συνεργασία στην έκθεση πρωτοβουλίας αυτής. Παρά τις αντιπαλόμενες απόψεις, καταφέραμε να βρούμε συμβιβασμούς. Και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των κουνελιών στην εκτροφή θεωρώ ότι είναι ένα, μια επιτυχία, γιατί επί 60 χρόνια δεν ήταν στην ημερήσια τέταξη της Επιτροπής μας το θέμα των κουνελιών. Και έτσι λοιπόν είναι σαφές ε, ότι εντοπίσαμε ποια είναι τα προβλήματα και θεωρώ ότι δίνουμε ένα μέλλον για την εκτροφή κουνελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα η έγκριση του κειμένου για την καθορισμό ελάχιστων προτύπων για την εκτροφή κουνελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συναδελφοί, είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε στην ολόνα και μεγαλύτερη επιθυμία για υψηλή ποιότητα προϊόντα, αλλά παράλληλα και για περισσότερη προστασία των ζώων. Και θα έπρεπε να θερούμε επιτακτική ανάγκη το να φροντίζουμε τους απροστάτευτους και να μειώνουμε τον πόνο που υπόκειται. Με κάποιες ελάχιστες εξαιρέξεις, σήμερα τα κουνέλια τα μεταχειριζόμαστε σαν αντικείμενα, χωρίς ζωή. Στις εποχές λοιπόν των μεγάλων αλλαγών τις οποίες διανύουμε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς τα έξω, προς τους πολίτες, προς τον κόσμο, ότι το κοινοβουλίο μας είναι κάτι παραπάνω από ένα ψυχρό ίδρυμα και ότι ακούμε και την καρδιά μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε καρδιά και τα χρησιμοποιούμε και για τα ζώα. Και θα σας ε, παρακαλούσα λοιπόν να εγκρίνετε την έκθεση και ιδιαίτερως την παράγραφο 16β με την αναφορά για τον καθορισμό στο μέλλον ελάχιστων προτύπων. Όλος ο πληθυσμός των κουνελιών θα σας ευγνωμονεί και σίγουρα και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Οι περισσότεροι από εμά, όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε κουνέλια στα σπίτια μας. Δεν είναι και τόσο περίεργο. Εγώ, ε, μάλιστα, άρχισα ε, θυμάμαι ότι είχα αρχίσει να κλαίω όταν σκοτώσαν το κουνελάκι μου παιδί. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε τους ε, συμβιβασμούς ηλεκτρονικά, ως συνήθως, και, το υπόλοι... και τα... τις υπόλοιπες προφορίες θα τις ε, ψηφίσουμε με ως χειρός. Ξεκινάμε ε, με το συμβασμό Α. Ψηφίζουμε. Πέραση της προφορίας. Έχουμε έναν υπεράριθμο ευρωβουλευτή από το ΕΛΚΑ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε εν συνεχεία στο συμβασμό Β. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της 82 παρακαλώ. Όχι, καταπίπτει αυτή η τροπολογία. Πάμε λοιπόν στον συμβασμό C. Ψηφίζουμε το συμβασμό C τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός D. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό D. Λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Θα ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 105, γιατί δεν είμαστε σίγουροι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 107. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε. Συμβασμός ε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική ε. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός έφα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός G. Ψηφίζουμε τώρα την συμβαστική G. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός H. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I. Ψηφίζουμε το συμβασμό I. Πέρας. Εγκρίνεται. 159. Τροπολογία 159. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 246. Ψήφι υπέρ. Της 246. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. Ελέγχουμε ξανά την τροπολογία 171 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 172 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβασμός K. τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση L. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία M. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβαστική τροπολογία ου 1, όμικρον 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την όμικρον 1. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον 2. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την συμβαστική τροπολογία όμικρον 2, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 213. Καταπίπτει όμως. Συμβαστική τροπολογία π. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 227. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 227. Πέρας τροπολογίας. Εγκρίνεται. Με τρεις ψήφους παραπάνω. Συμβαστική Q. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβαστική R. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Γκρίνεται. Τροπολογία. Όχι. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 2.32. Συμβαστική τροπολογία S. Πέρας. εγκρίνεται. 243. Ψηφίζουμε την 243. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 243 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Με μόλις μια ψήφο παραπάνω υπέρ. Συμβαστική τροπολογία τι. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 252. Καταπίπτει, κάνω λάθος. Και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ εγκρίνεται 5 υπέρ εγκρίνεται 6 υπέρ εγκρίνεται 7 υπέρ εγκρίνεται 8 υπέρ εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Ζαμικό Πέρασε τροπολογία της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 17 λοιπόν. Άρα 11. Ψηφίζουμε την 11. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της 11. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 2. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Τώρα εντάξει, αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Ωραία. Επανερχόμαστε λοιπόν στη συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 40. Νομίζω ότι καταπίπτει. Ναι, πράγματι. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία επί τη συμβαστικής 5. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 6 πέρας εγκρίνεται συμβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 66 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 69 Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί βλέπω ότι ίσως η πλειοψηφία είναι η ίδια. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. 70. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Και στη συνέχεια 71 παρακαλώ υπέρ εγκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να περάσουμε να ψηφίσουμε το σχέδιο όπως έχει τροποποιηθεί. Δεν βλέπω αντιρρήσεις ή σχόλια, προτάσεις, άρα άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η πρόταση και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Εκ. Μήπως θα ήθελε να πάρει το λόγο μετά την ε, ψήφιση, αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πετύχαμε μια συμφωνία για ε, πολλά ζητήματα και Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι τελικά δημιουργήσαμε μια τίγρη χωρίς δόντια. Μια πρωτοβουλία δηλαδή, η οποία θα περάσει στην Ολομέλη στη συνέχεια στην Κομισιό. Αλλά δεν θα περιλαμβάνει καμία μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία από νομοθετή τη άποψη. Τι νόημα έχει. Ωραίο παιχνιδάκι. Ωραίο παιχνιδάκι για να ησυχάσει και να καθησυχάσει τη συνείδηση των μισών ευρωβουλευτών. Αλλά δυστυχώς δεν θα βοηθήσει τα ζώα που υποφέρουν, που πάσχουν. Εγώ σας το λέω, δεν μπορώ και να υποταχτώ. Θα τα πούμε και πάλι στην Ολομέλεια με μια τροπολογία η οποία θα περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το απόσπασμα το οποίο βγάλαμε εδώ και θα α, παλέψουμε νύχια και με δόντια. Δεν το λέω επιμορφή απειλής, το λέω επιμορφή υπόσχεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο γιατί ότι ο συνάδελφος Πόλτσακ, ο οποίος ε, ε ήταν υπεύθυνος εκ ονόματος της ομάδας έχει φύγει από την Επιτροπή πλέον. Είναι μεν παρόν εδώ σήμερα και θα θέλω να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκανε για την ομάδα μας και την Επιτροπή μας. Ο Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία τον εισηγητή. Θα μας λείψετε και καθόλου δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση που λάβατε είστε τόσο νέος, ε, έχετε μέλλον και μπορεί να επανέλθετε κάποια στιγμή στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε και ελπίζω να το ξαναπούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή πάλι. Δεν σημειώσαμε πρώτα κατά 100% αλλά νομίζω ότι πρόκειται για ένα καλό βήμα σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και να περάσουμε στο 12 της ημερήσιας διάταξης. Για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και φροντίδα των υποειδών. Και υπεύθυνη η συγκεκριμένη είναι η κυρία Γκέρλινγκ ε, Τζούλη. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο, εφόσον είναι στην αίθουσα. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μιλάω με κάποιο δισταγμό, γιατί ε, δεν θέλω να μην σα ε, προκαλέσω και σε κίνηση. Δεν φαντάζομαι να είχατε και υποειδές το οποίο να πέθανε. Αν ε, είχατε όμω θα βρείτε πολλέ λεπτομέρειε εδώ πέρα στην έκθεσή μα για το πώ θα βελτιώσουμε τη μεταχείριση των ζώων αυτών, γιατί οι άνθρωποι και τα ζώα είναι φίλοι εδώ και και με το κείμενο αυτό βελτιώνουμε τη φροντίδα των ζώων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω λοιπόν στην ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κα... Υπέρ. Κα... Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Απαρρίπτεται. Η 3. Υπέρ. Κα... Εγκρίνεται. Η 4. Υπέρ. Εγκρίθηκε. πέντε Υπέρ. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική α. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ναι, όντως, συμβαστική α ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική β. Έναξη. Ψηφοφορία για τη συμβαστική β. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στη συμβαστική ηθή. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική D. Ψηφίζουμε τη συμβαστική D. Πέρασε. 118. 118. Ε, τροπολογία 118. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Εγκρίθηκε. 120. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε για σιγουριά. Την 120. Την 120. Παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για επαλήθευση. Περάσει. Και δεν είμαι σίγουρος ότι σηκώσατε καλά τα χέρια σας. Συμβαστική ε. Έναρξη ψηφοφορίας για την ε. Πέρες. Εκατόν Κύριε Σαραμπέλα. Και καλωσορίζω και τον κύριο Τραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. G, παρακαλώ. Γιατί την G. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 228. 228 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 228. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω τον κύριο Ντόρφμαν. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική H. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΆΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν εξήντα έξι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Α, όχι, με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική L. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και πάλι εγκρίνεται. Συμβαστική M. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 219. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 220. του κυρίου Αρτουή. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε καλύτερα. 220 αρχίζει η ψηφοφορία. Κύριε Καϊνόφσκι, νομίζω ότι κάνατε λάθος. Πέρας. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 227 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. Συμβαστική ο όμικρον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 232 υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Συμβαστική π. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και πάλι εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική R. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική S. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τι, ταφ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95 του κυρίου Καπούτο, υπέρ. Εγκρίνεται. ...204, τροπολογία 204, που είναι ίδια με τη 251, υπέρ. Εγκρίνονται. Συμβαστική U, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και πάλι εγκρίνεται. Συμβαστική VA. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 9. Τροπολογία 9 της εισηγήτριας ΠΕΡ. Εγκρίνεται. W. Συμβαστική W αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική X αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Y, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην Z. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την 33. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 37. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική διπλό α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική διπλό β. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέρας ε, της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κύριο Χάιτεμαν υπέρ κατά ας ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται Διπλό δέλτα, συμβαστική, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Διπλό ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Διπλό F, συμβιβαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εβδομήντα δύο υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο στο σύνολό του, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του σχεδίου έκθεσης. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε κυρία Γκέρλινγκ το λόγο για να μας πείτε κάτι. Φαίνεται πως όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Νιου. Ένα σημείο για τη ιστορική σημασία, Πρόεδρε. Για τα πρώτα 7,5 χρόνια πέρασε μία τροπολογία γνώση αυτή την Επιτροπή. Είτε αποφασίσατε να είστε ευγενεί μαζί μου επειδή νομίζατε ότι έχω τα γενέθλιά μου, είτε σιγά σιγά σας μετακινώ στο σωστό δρόμο. Why did you vote against the report? Γιατί καταψηφίσατε την έκθεση τότε. Είναι απίστευτο. Με ρώτησαν γιατί καταψήφισα την έκθεση. Πάντα είναι πολιτική του UKIP να ψηφίζει κατά των εκθέσεων. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα περάσουν αυτά τα πράγματα, πολύ απλά προσπαθούμε να περάσουμε κάποιες καλές τροπολογίες. Αυτό είναι το σύστημά μας και αυτό ακολουθώ πάντα. Bravo pana ε, και έχετε δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η δημοκρατία άλλωστε. Αυτό επιτάσσει. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διατάξη σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για το 2015 Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Γιάχα. Από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και ο κύριος Σέλερ θα είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Ο κύριος Γιάρ φαντάζομαι θα θέλει να πάρει το λόγο από αυτό. Να μην σας θερήσω την ευκαιρία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους και οδησυσυγητές συμβιβαστικέ τροπολογίε ε, καταφέραμε να βρούμε που καλύπτουν 36 τροπολογίε και χαίρομαι ιδιαίτερω. γιατί η συνεργασία των ε, σκιωδών ήταν εξαιρετική και δεν επηρεάστηκε από τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πραγματικά Πολύ καλή συνεργασία και αυτό φαίνεται στην έκθεση, πιστεύω. Για το περιεχόμενο τώρα, για τη χορηγήση απαλλαγή. Διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό σφάλματος ε, μειώθηκε κατά 2,9% στο γεωργικό τομέα. 2,2 είναι ε, στον πρώτο πυλώνα η απορρόφηση. Αυτό είναι αρνητικό. Και στην έκθεση Ζητήσαμε και εφαρμόσαμε καλύτερο διαχωρισμό των ειδών σφαλμάτων. Υπάρχουν τα σφάλματα που δεν έχουν και οικονομική επίπτωση και αυτά φυσικά θα πρέπει να διακρίνονται από αυτά που προκαλούν πολιτική και οικονομική ζημιά, που έχουν οικονομικές συνέπειες. Και έχουμε και την Γενική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη για το 2015, την ορίσαμε. Και το θέμα αυτό φυσικά επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ε, γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο της λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι πολύ ευτυχής η συγκυρία της έκθεσης και για τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Καταφέραμε λοιπόν ε, τα χρήματα τα οποία, τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μα, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, να χαμηλότερο ποσοστό σφάλματο. Άρα προβλέπω στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στον κανονισμό και στη γνωμοδότηση. Εάν ε, το επιθυμείτε, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψήφιση της, τροπο, ε, της συμβαστικής τροπολογίας F. Ψηφίζουμε. Το πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ψήφι ΠΕΡ, Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. 12 υπέρ εγκρίνεται 15 υπέρ εγκρίνεται 14 υπέρ κατά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά το σημείο αυτό Τροπολογία 14 δηλαδή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Το περιμένω ψηφίσει κυρία Νόιχερ. πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Α. Ψηφίζουμε εικονικά πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική Δ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Τσι. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 42. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 και 44 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ελέγξουμε ευθυνικά αυτές τις δύο. 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σαράντα επτά υπέρ. Σαράντα εννιά υπέρ. 46. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Ψηφίζουμε την 59 αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε απορρίψει την 50. Ποιο είναι υπέρ τη 59, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 51 του κύριου Γιάρη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική C. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Του κύριο Σόνι. Ψήφι ΠΕΡ. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 67. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Μπράβο κύριε Σάνι. Για μία ψήφο. 71. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ της 73. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ψηφοφορία, την τελική του σχεδίου γνωμοδότησης με τις τροπολογίες. Ψηφίζουμε τώρα. ο ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θέλει να πάρει το λόγο ο εισηγητής. Όχι. Τότε να πω εγώ συγχαρητήρια και για την παρουσίαση και για την έκθεση. Τελειώσαμε λοιπόν τις προφορίες. Και περνάμε τώρα στο σημείο 14. Μάλιστα δεν έχουμε καθυστερήσει καθόλου το αντίθετο. Ξεκινάμε νωρίτερα το επόμενο σημείο. Ο κύριος Γέγας είναι εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε στο σημείο 14. Ο σωστό συνδυασμό χρηματοδότηση για τι περιφέρειες τη Ευρώπη, ισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια νέα ιδέα. Θέλουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, με πιο αντικειμενικό τρόπο και με καλύτερο τρόπο σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, έγινε μια διάσκεψη στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες, βέβαια, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης και βοήθειας προς περιφέρειες. Είναι μια γνωμοδότηση, έκθεση της Επιτροπής ΡΕΓΚΙ. Ο κ. Βιέγας την ετοίμασε, είναι ο συντάκτης. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας μιλήσει για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, για τις πιστώσεις, για εργαλεία μικροχρηματοδότησης, ε, εργαλεία ιδίων πόρων και ιδίων κεφαλαίων που αντικαθιστούν τις επιχορηγήσεις. Κύριε Βιέγας, έχετε την, το λόγο για να παρουσιάσετε το κείμενό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις αυτών των ε, χρηματοοικονομικών μέσων σε επίπεδο γεωργίας. Κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης ή γνωμοδότησης πραγματοποίησαμε δύο ακροάσεις, μία στην Πορτογαλία και την άλλη εδώ στο Κοινοβούλιο, όπου καλέσαμε τις οργανώσεις και ε, αγροτικές ενώσεις για να δούμε τι επιθυμούν. Και το κείμενο αυτό είναι απότοκο αυτής της συνεισφοράς των αγροτικών οργανώσεων που θέλησαν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση αυτού του σχεδίου και μας έστειλαν και στοιχεία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη συνέχεια μετά από τις ακροάσεις. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας γνώμη. Ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, αυτό που μας απασχολεί είναι ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την κατάσταση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτούς τους μικροπαραγωγούς πρωτίστως. Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς στα πλαίσια της ΚΑΠ και βλέπουμε ότι πολύ λίγες είναι εκείνες οι χώρες που ενέταξαν τα χρηματοδοτικά μέσα στα ε, προγράμματα περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, από αυτά που βλέπουμε και διαπιστώνουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα μέσα έχουν μία δυναμική. Γιατί σε επίπεδο γεωργίας βλέπουμε κρίσιμα σημεία που έχουν σχέση με την πρόσβαση στο πιστοδοτικό σύστημα. Και διαγράφονται πολλές δυνατότητες βάσει αυτών των μέσων. σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις που λαμβάνουμε, υπάρχει ομοφωνία ότι τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Δεν θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν. Αυτό μας λέει ο αγροτικός κόσμος. βεβαίως αναγνωρίσουμε τη δυναμική πορεία αυτών των χρηματοδοτικών μέσων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μεγάλες υποδομές, τις αρρώσιμες γές, τις μεταφορές, ένα συσχετισμό δηλαδή στοιχείων που θα μπορούσαν να τύχουν της υποστήριξης ε, παρομοίων μέσων χρηματοδοτικών μέσων. Γνωρίζετε το κείμενο και θα, θέλαμε, θα ήθελα τώρα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ήταν πολύ σύντομος. Έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και την εισηγητή για την πρόταση αυτή και για την εισαγωγή που μας έκανε. Είμαι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα μιλήσω λοιπόν για την έκθεση αυτή και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο και κέριο το θέμα αυτό. Σήμερα δεν μπορούμε να ζούμε σε απομόνωση. Ο αγρότης περιτριγυρίζεται από μια κοινωνική δομή, ένα κοινωνικό ιστό. Χρειάζεται εκπαίδευση, κοινωνικέ υπηρεσίε, αυτό και η οικογένειά του. Υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμικέ υπηρεσίε. Το πρόγραμμα Leader που ασχολείται με τον δεύτερο πυλώνα έχει ως σκοπό όχι μόνο τη γεωργία, αλλά και τι ε, γεωργικές επιχειρήσεις, τι δημόσιες υποδομές, για τη βελτίωση της συνεκτικότητας της ζωής των αγροτών. Μία δανεική λύση θα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα περιφερειακά, τα, τα ταμεία συνοχής και τα τριφαντικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό οι αγρότες θα μπορούσαν να λάβουν από κοινού αποφάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ε, ταμείων στην κάθε περιοχή. Αυτό θα βοηθούσε να αναπτυχθούν πιο γρήγορα οι περιφέρειες. Γιατί συνήθως όταν οι επιχειρήσεις ε, αναπτύσσονται γρήγορα, δεν θα έχουν ευκαιρίε να αναπτύσσονται γρήγορα οι επιχειρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Λιθουανία, κάνουν λάθος λάθος όταν τα χρήματα που ωφελούν αυτές τις κοινότητες και τους αγρότες ε, τελικά για τις ε, χορηγήσεις αυτές τις, ε, τα χρήματα αυτά καρπώνται το όφελος το πολιτικό το κέντρο της χώρας και ουσιαστικά αποδυναμώνονται οι περιφέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία πρόταση ζητώντας από τα κράτη-μέλη να αφήσουν στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο την ε, πρόσθετη αυτή αξία των διορθωτικών ταμείων, των ταμείων συνοχής, των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι, οι περιφέρειες μπορούν να ωφεληθούν άμεσα, να μην αφήσουμε δηλαδή να περάσουν όλα αυτά σε κεντρικό επίπεδο. Αυτή θα ήταν η πρόταση μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις επεξηγήσεις. Το θέμα αυτό είναι ύψης της σημασίας ως προς την χρήση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τον αγροτικό κόσμο. Εγώ είμαι ε, αναπληρωματικό μέλος στη Ρέτζη και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στην απορρόφηση, γι' αυτό χρειάζεται συνέργεια μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευφυής όπου οι άνθρωποι να ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υποδομές. Αυτό αφορά το σύστημα υγείας, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη χρήση του διαδικτύου και ούτω καθεξής. Εάν δεν γίνει δελεαστικός, δελεαστική ύπεθρος, δεν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους μικροπαραγωγούς στην Ήπεθρο. Εγώ ως κοιόδης θα υποβάλω τροπολογίες για τον συνδυασμό αυτών των χρηματοδοτικών μέσων για να φτάσουμε και με τη χρήση του ορίζοντα 2020, το ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία σε ένα ενίο πλαίσιο δράσης. Θα πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία προσέλκυσης των αγροτών. Να τους δώσουμε νέες ευκαιρίες έτσι ώστε να μπορούν να καρποθούν αυτό το πλαίσιο και να μπορέσουν ε, να δράσουν. Γνωρίζουμε ότι το πιο δύσκολο είναι όχι η παραγωγή, αλλά η μεταπόληση της παραγωγής. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτό το δίκτυο μεταπόλησης των προϊόντων που διαθέτουν οι αγρότες. Έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας της Βραζιλίας μας μίλησε για αυτό το πλαίσιο της αποδοτικής και ανταγωνιστικής γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και να πω και εγώ δύο κουβέντες. στην πολιτική συνοχή είναι σημαντικό τα χρήματα να πηγαίνουν πραγματικά στις χώρες που τα χρειάζονται. Γιατί θυμάμαι όταν ε, ήμουν στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, το τόνιζα σε αυτό. Η πολιτική συνοχή λοιπόν θα πρέπει να τα λάβει υπόψη αυτό και το ξέρω ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή, συχνά αναφέρονται ότι υπάρχει ο δεύτερο πυλώνα. Αλλά ο δεύτερο πυλώνα δεν ωφελεί πάντα τον σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορώ να πάρω το λόγο για την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ στο σημείο 4. Πολλά αναφέρονται στην έκθεση και σίγουρα είναι σωστά και όλοι γνέφουν καταφατικά και συμφωνούν, αλλά το θέμα είναι στο σημείο 4, όπου ξεκαθαρίζεται ότι όλα όσα μπαίνουν στο δεύτερο πυλώνα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι εις βάρος στο πρώτο πυλώνα. Όλοι ξέρουμε ότι αν κάνουμε πιο πολλά για το δεύτερο πυλώνα και είμαι υπέρ, 100% υπέρ της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, αλλά το ξέρω ότι αυτό ενδεχομένως είναι εις βάρος του πρώτου πυλώνα, αν παραμένει καν αυτό το μοντέλο και εξακολουθήσει να υπάρχει. Και νομίζω ότι για λόγους τιμιότητα και εντιμότητας θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα, δεν λέμε να χτυπώσουμε και τα χρήματα. Εννοούμε ότι θα πάρουμε από κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Από άλλου τομεί. Δεν θα έρθουν φρέσκο χρήμα Άρα ουσιαστικά να πούμε τίμια ότι τα χρήματα αυτά θα φύγουν από τον πρώτο πυλώνα και όλοι όσοι α, ε, χειροκροτούν και είναι ικανοποιημένοι απλά να το πούν τίμια. Είμαι υπέρ του να μεταφερθούν χρήματα από τον πρώτο πυλώνα για έργα τα οποία έχουν νόημα και βγάζουν νόημα. Απλά να το πούμε ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Oui, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το σημείο Β. Περιγράφει την ε, οικογενειακή γεωργία όπως, ως παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής και εγγυητή της ε, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της γεωργίας μας. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό, γιατί το μέγεθος των ε, εκμεταλλεύσεων στην πραγματικότητα και αυξάνεται. Και στη Γαλλία, μάλιστα, έχουμε ένα σύστημα εξαφάνισης πολλών μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ε, και τελικά αυτό το μοντέλο προωθεί τι ε, μεγάλε ε, βιομηχανικού τύπου εκμεταλλεύσει. Επίση το σύστημα 4. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε την, το σύστημα χρηματοδότηση να αντικαταστήσει τι χορηγήσει. Η ιδιωτική χρηματοδότηση όλο και μεγαλώνει και αυτό μεγαλώνει την εξάρτηση των γεωργών από τι τράπεζε, οι οποίοι εξαγείρονται εναντίον αυτού. εξαρτούνται απόλυτα, ας πούμε, και πιέζονται πάρα πολύ από τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει, να αντιδράσει σε αυτό. Γιατί ε, τα διάφορα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότηση, ε, το FEDER, το FEADER για την περιφέρειά μου, δεν κατάφεραν να, να αντισταθμίσουν τι εδαφικέ ανισότητε. Το ερώτημα είναι, με ποιο τρόπο θα διευκολύνετε λοιπόν τι επενδύσει, χωρί να παραδώσετε το γεωργό στην πίεση, α πούμε, των τραπεζών που θέλουν να αποπληρωθούν τα δάνεια που, δίνονται, που δίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση. Είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Παραμονή της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού, δημοσιονομικού πλαισίου. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να οδηγήσει σε βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώ πιστεύω ότι εμεί τα μέλη τη Ευρωπαϊκή ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Γεωργίας θα πρέπει να θεωρούσουμε τη Γεωργία ως ένα πολυεπίπεδο τομέα και μέσα από τα πολλαπλά εργαλεία της, ε, πολιτική της πολιτικής θα πρέπει να την προωθήσουμε. Θα πρέπει, πιστεύω, να προωθήσουν αυτά τα εργαλεία την περιφερειακή ανάπτυξη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει όμως να είναι ο μόνος τρόπος ε, οικονομικής ε, υποστήριξης και χρηματοδότησης. Οι γεωργικές περιφέρειες είναι μακριά από τα κέντρα συνήθω, τα διοικητικά κέντρα κτλ. Και αυτό καθιστά το πρόβλημα των υποδομών πολύ πιο οξύ και φυσικών υποδομών και οικονομικών υποδομών, Γι' αυτό στην τελική μορφή της έκθεσης θα πρέπει να τονίσουμε την απόσταση αυτή που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές και τα κέντρα διοικητικά και άλλα. Και όταν χρησιμοποιούμε οικονομικά εργαλεία θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε συλλογικά προγράμματα που προωθούν τις τοπικές πρωτοβουλίες και την ταυτότητα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε του κλειστού κύκλου παραγωγής. Και γιατί το λέω αυτό. Μέσω των επενδύσεων σε κλειστούς κύκλους υποστηρίζουμε και τις πρώτε ύλε, οι περισσότερε εκ των οποίων προέρχονται από την εν περιφέρεια, καθώς και στην, την επεξεργασία, ε, συσκευασία και αποθεματοποίηση που γίνονται στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε και το εργατικό δυναμικό στην συγκεκριμένη περιοχή, αναστρέφουμε την τάση απομάκρυσης του πληθυσμού, γιατί η αστιφιλία είναι μέγιστο πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο όμως τονίζουμε την τοπική οικονομία και την κάνουμε λιγότερο εξαρτημένη από το κέντρο. Έχω και άλλες προτάσεις, αλλά θα σας τις παρουσιάσω γραπτώς ως τροπολογία στο σχέδιο γνωμοδότησης πιστεύω ότι όλοι στο ίδιο μήκο ε, κύματο ε, βρισκόμαστε, άρα θα πρέπει οι μένα υποστηρίξουν του δε. Πολύ ωραία, κύριε κ. Τόρφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πώς καταλαβαίνω το σημείο 4. Δεν συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Νόχιλη, συνάδελφος. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι η συζήτηση μεταξύ πρώτου και τέσσερου πυλώνα. Νομίζω ότι το θέμα είναι κατά πόσον θέλουμε επιδοτήσεις στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα ή θέλουμε χρηματοοικονομικά μέσα. Γι' αυτό νομίζω ότι το σημείο 4 που περιλαμβάνεται σε σχέση με τις επιδοτήσεις ε, δεν θα πρέπει να μειώσουν τα ταμεία αυτά και τις επιδοτήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε για τη διατήρηση των ε, χρηματοοικονομικών μέσων. Γιατί σε εποχές όπου είναι πολύ μοντέρνα τα εργαλεία και τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως το ΕΦΣΥ, υπάρχει τάση να μειώνουν τις επιδοτήσεις. Δεν συμφωνώ στο σημείο 5, επίσης. να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στα κοινωτικά προγράμματα ή τα χρηματοοικονομικά μέσα. Κοιτώντα, α πούμε, το ταμείο του Juncker, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται να υπάρχουν πλατφόρμες τις οποίες να χρησιμοποιούν οι μεμονωμένοι αγρότες και εκτροφείς. Για παράδειγμα, η Νέε επιχειρήσει οι νεαροί αγρότε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι επί τη αρχή τέτοιε πλατφόρμε χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από μεμονωμένε επιχειρήσει. Επόμενος. Ευχαριστώ. Είμαι από την Επιτροπή προπολογισμού. Συμμετέχω και στην Επιτροπή Προπολογισμού. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο ε, χρησιμοποιείται στον προπολογισμό εκτό ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια διευκόλυνση η οποία όμως θα προκαλέσει προβλήματα γιατί στα χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι είμαι κατά όλων ε, αυτών των μέσων, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Όχι να ξεχνάμε τις επιδοτήσεις σε κάποιες τομείς της πολιτικής λόγω των τεχνικών μέσων, όπως είναι η αγροτική πολιτική, η πολιτική για την υπεθρο. Άρα, πιστεύω ακράδαντα ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα κάτσουμε να σκεφτούμε σωστά. Όλα τα αγροτικά ταμεία, όχι μόνο τα γεωργικά ταμεία, όχι μόνο η ΚΑΠ και ο δεύτερος πυλώνας, αλλά και άλλα ταμεία. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα χρηματοοικονομικά μέσα. Άρα, εγώ είμαι πολύ διστακτικό για τα χρηματοοικονομικά μέσα και ελπίζω να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα στεναρό οικοδόμημα για την ΚΑΠ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα θέλει το λόγο να... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, συγγνώμη. Δεν έχω στον κατάλογο το όνομά σας. Λυπάμαι πολύ. Yeah, good afternoon. Thank you, Chairman. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρο Μιχαήλ Πιούκερ από την DG uh, ε, Γεωργίας. Ooh. Ε, ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Να καλωσορίσουμε το σχέδιο χρηματοδότηση τη Επιτροπή ε, σα για την ε, ανάπτυξη και το δυναμικό τη γεωργία στι γεωργικέ περιοχέ και στην Υπεθρό. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα εργαλεία αυτά, τα μέσα αυτά, είναι συμπληρωματικά προ τι επιδοτήσει. Και φυσικά σε θέματα επιδοτήσεων στη Γεωργία και στην ανάπτυξη της πέτρου έχουμε πιο πολλή εμπειρία. Αλλά από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια ανάγκη που υπάρχουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στις αγροτικές περιοχές. Με τις επιδοτήσεις έχουμε φτάσει στα όρια μας. Έχουμε κάποιες αιτήσει όπου λαμβάνουμε υπερβολικέ αιτήσει και πολλοί γεωργοί και αγρότε δεν λαμβάνουν τι επιδοτήσεις αυτέ. Ή σε άλλε καταστάσει βλέπουμε γεωργού που δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση γιατί ο οικονομικός κλάδος διστάζει να χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα, μικρές επιχειρήσεις. Άρα θεωρούμε ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούν ένα τέλειο εργαλείο για να συμπληρώσουμε αυτά που εφαρμόζουμε έτσι κι αλλιώς στην πολιτική μας για την ανάπτυξη της Πέτρου. Σε ό,τι αφορά το συμπληρωματικό χαρακτήρα, λοιπόν. Δεν εφαρμόζουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα έτσι απλά, από ό,τι ξέρετε. Τα κρατή μέλη που θέλουν να εισαγάγουν στο πρόγραμμα ανάπτυξη πέτρου ένα χρηματοοικονομικό μέσο, χρειάζεται να κάνουν μια εξάντε αξιολόγηση πριν τα χρησιμοποιήσουν. Και αυτό χρειάζεται ακριβώ για να εγγυηθεί αυτό ο συμπληρωματικό χαρακτήρα. Γιατί αν δεν υπάρχει πραγματική πρόσβαση στο κεφάλαιο ή ανάγκη ή κενό για την πρόσβαση στο κεφάλαιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη του χρηματοοικονομικού μέσου. Και έτσι λοιπόν εξασφαλίζεται αυτή η προδιαγραφή. Από την άλλη, τα χρηματοοικονομικά μέσα δίνουν επιπρόσθετο δυναμικό σε νέους, για παράδειγμα, και οργούς. Χρηματοδότηση η οποία δεν είναι δυνατή υπό άλλα συστήματα. Είναι σημαντικό όμως όσο ξεκινάνε την για τους που ξεκινάνε μια επιχείρηση. Από πλευρά της Επιτροπής λοιπόν τι κάνουμε προωθούμε με προσοχή τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά με τρόπο που αξιολογούμε πραγματικά με τα κρατημέλη την ανάγκη για το χρηματοοικονομικό μέσο. Παρέχουμε συγκεκριμένο και στοχευμένο coaching και παροχή συμβουλών. Και κοιτάμε τις ανάγκες, τις συγκεκριμένες ανάγκες του κράτους μέλους δεν έχουμε μία λύση κομμένη και ραμμένη για όλου. Εξετάζουμε τι διαφορέ που υπάρχουν από κράτο μέλο σε κράτο μέλο ιδιαίτερω. Συνοψίζοντα, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε μεν το σχέδιο έκθεσης, αλλά σα καλούμε και εσάς να προωθήσετε τα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να εκφραστεί η ανάγκη τόνωσης των μέσων αυτών, γιατί τουλάχιστον θεωρούμε ότι πρέπει να δοκιμαστούν τα μέσα αυτά, Συμπληρωματικό πώ. Αλλά χαιρόμαστε που είτε οι 49 αρχές κάνουν σχετική αξιολόγηση για να δουν κατά πόσον το μέσο αυτό θα είχε νόημα να εισαχθεί στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης της Πέτρου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάνεγκαν, θέλετε το λόγο. Ναι, πράγματι, θα ήθελα να πω και να καταγραφεί ότι τα χρηματοδοτικά ε, μέσα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις άμεσες πληρωμές γιατί αυτό με ανησυχεί και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ε, έρευνα σε σχέση με το χρέος των αγροτών και φοβάμαι ότι θα γίνουν ακόμα πιο, ε, θα εξαρτώνται ακόμα περισσότερο από τις δανειοδοτήσεις. Και θα ήθελα να πω ότι έχουμε την παλιά ιστορία που ακούμε και από τους αριστερούς. Εάν οι αγρότες πραγματικά κέρδισαν από την παραγωγή τους και είχαν και ένα μεγάλο και είχαν και ένα κέρδος, τότε δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό δεν μπορούμε τεχνητά να δημιουργήσουμε τιμές για κάποιον ο οποίος ε, αποβλέπει στο κέρδος. Εάν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική θα εξακολουθούμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Βιέγκας, έχετε το λόγο ως εισηγητής. Εντάχει, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει συνένεση σε σχέση με το ζήτημα αυτό για να υπάρχει ένα συμπληρωματικός χαρακτήρας αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Ακούστηκαν πολύ σημαντικές ιδέες που θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να εντάξουμε στο κείμενο, το οποίο δεν πρέπει να είναι και πολύ εκτενές, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτών που ζουν στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ευρύ φάσμα ε, υποστήριξης που έχουμε στη διάθεσή μας, μέσων στήριξης δηλαδή, και θεωρώ ότι οι επιδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε το εισόδημα των αγροτών που προέρχεται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Εδώ μιλάμε για το πρώτο πυλώνα. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δίκτυα που χρησιμοποιούν για να προωθήσουν την παραγωγή τους και νομίζω ότι θα πρέπει να, δούμε τις κατάλληλες, να βρούμε τις κατάλληλες υποδομές για να αυξήσουμε την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Και ως προς το σημείο 5 φαίνεται ότι αποκλείεται η ατομική χρηματοδότηση, οι μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις, κάτι το οποίο δεν θα δεχτούμε ούτε και στο κείμενο. Εγώ καταγράφω αυτή την ευρεία συνένεση και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσω να δεχτώ τις υποδείξεις σας και θα φτάσουμε σε ένα συνενετικό κείμενο όπου ο καθένας θα αναγνωρίζεται, θα αναγνωρίζει τα δικά του δεδομένα σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Βιέγκας. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ε, είναι η 26 η Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Χαίρομαι γιατί μπορέσαμε και προχωρήσαμε με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που υπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς μας, δηλαδή μπορούμε να στηρίξουμε ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό αγροτών. Η, την απόφαση βεβαίως την ε, παίρνουν οι τράπεζες κατά μείζωνα λόγο. Μιλάμε για επιχορηγήσεις και όχι μορφές ε, άμεσων πληρωμών. Μιλάμε λοιπόν για επιχορηγήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις άμεσες πληρωμές. Και βεβαίως τη στιγμή που ζητάμε τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα ήταν ε, πραγματικά πολύ επίκαιρα και ενημερωμένα. Περνάμε στο σημείο 15, ε, βιολογική παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων και τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι ε, μια έκθεση που έχει αναλάβει ο κύριος Χόισλινγκ έγινε μία ενημέρωση για, τις, ε, για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Είχαμε 14 ε, τριμερείς μέχρι τώρα και φαίνεται ότι προσεγγίζουν ε, τις θέσεις τους τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά η Σλοβακική Προεδρία δεν έδωσε τελική μορφή σε αυτές τις, σε αυτές τις θέσεις γιατί υπήρχαν διχογνωμίες. Θα θέλαμε ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Μάλτας να μας μιλήσει επί των εξελίξεων, αλλά θα δώσουμε καταρχήν το λόγο στον κύριο Χόισλινγκ για να μας πει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι τριμερείς και κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες ολοκλήρωσης. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, το θέμα αυτό το έχω αναλάβει αρκετά συχνά. Και ελπίζαμε να σημειώσουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σύντομα, να ευχαριστήσω και τη Σλοβακική Προεδρία για το ότι όντω σημειώθηκε πρόεδρο σε πολλά σημεία και υπήρξε προσπάθεια να πετύχει και μια τελική συμφωνία η Σλοβακική Προεδρία. αλλά ο συμβιβασμό δεν βρήκε σύμφωνο ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο. Και τελικά δεν υπήρχε λοιπόν συμφωνία πέρσι. Και έτσι τώρα το ανέλαβε η Μαλτέζικη Προεδρία. Να αναφέρω τα τέσσερα σημεία για τα οποία δεν υπήρξε συμφωνία. Το θέμα των ε, φυτουρίων, το θέμα του τερματισμού των ε, εξαιρέσεων, το θέμα των ε, προληπτικών μέτρων ή τα όρια για τα φυτοφάρμακα και τέταρτον οι σπόροι. Αλλά ούτε στους βελτιωμένους ελέγχους μακροπρόθεσμα δεν πετύχαμε συμφωνία και εδώ υπάρχει θέμα στην εφαρμογή. Από πλευρά του Κοινοβουλίου δείξαμε μεγάλη διάθεση συμβιβασμού στις τελευταίες συνεδριάσεις, στους τελευταίους ε, τρομερείς διάλογους. το θέμα, για παράδειγμα, των κοινών ε, επεξεργασιών, για παράδειγμα, και σε πολλά άλλα σημεία όπου θεωρήσαμε ότι με μια επίδειξη καλή διάθεση θα κινητώνει και το Συμβούλιο λίγο. Αλλά δυστυχώ το Συμβούλιο πρέπει να ομολογήσω ότι από την πρώτη ε, διαπραγμάτευση δεν τροποποίησε καθόλου την εντολή του για τι διαπραγματεύσει και αυτό πάντα είναι δύσκολο για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε ότι όταν κάνουμε συμβιβασμού θα δεχτεί το αποτέλεσμα και το Συμβούλιο. Και έτσι δεν υπήρχε κοινιαία τοποθέτηση στους κόλπους του Συμβουλίου. Αντιθέτως, είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των ε, μελών του Συμβουλίου και θα δυσκολευτεί το άλλο το Συμβούλιο να βρει μια συμφωνία. Ελπίζουμε από μαλτέζικες πλευράς με την οποία ήδη έχουμε κάνει συζητήσεις θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια κοινή θέση των κρατών μελών. Και η Μαλτέζικη Προεδρία βρίσκεται σε φάση διεξαγωγής διμερών διαλόγων. Το νωρίτερο στα τέλη Μαρτίου θα τα πούμε στα πλαίσια του 10ου, του 5ου τριμερούς διαλόγου. Μετά το Δεκέμβριο και την αποτυχία του Δεκεμβρίου είπαμε ότι θέλαμε να κάνουμε μία παύση, μία διακοπή των διαπραγματεύσεων. Γιατί όλοι πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν κατά πόσο μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα όπω ω τώρα. Μπορεί στην τελική ανάλυση να μην καταφέρουμε καν να βρούμε μία συμφωνία. Αν τελικά ε, χρειαστεί να κάνουμε τόσους πολλούς συμβιβασμούς που τελικά δεν θα περάσει η θέση μας του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενδεχομένω δεν υπάρχει δυνατότητα εξέβρισης συμφωνία. Αυτό το λέμε με σαφήνεια. Και πολύ απλά δηλώνω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περιμένουμε κάποια αλλαγή, κάποια κίνηση, κάποια, ένα, κάποιο δείγμα καλή θέληση. Μπορεί να υπάρχει κάποια συμβαστική λύση, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να μπορούν να είναι και εφικτά στην πράξη. Συναμιλήσαμε και με, διάφορους, ε, με διάφορες ε, επιχειρήσεις, ε, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να θέσουμε οριακές τιμές, απλά θέλουμε μια έκθεση η οποία να αποτυπώνει στην πραγματική κατάσταση. Εμεί από πλευρά μα σα λέω, κάναμε συμβαστικέ προτάσει. Περιμένω κάτι τέτοιο και από το Συμβούλιο όμω πλέον. Και περιμένω και μια σωστή στάση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό με εκνεύρισε. Να σα πω την αλήθεια. Αυτό που με εκνευρίσε ήταν μια συνέντευξη του Επιτρόπου για τη Θεματογεωργία σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα, που ξαφνικά έβαλε ένα σύνδεσμο και δημιούργησε ένα σύνδεσμο μεταξύ ε, ασθένεια ασθένειας ε, και της ε, πολιτική και των ε, φυτοφαρμάκων. Και έκανε λοιπόν αυτόν τον αυθαίρετο σύνδεσμο. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Δεν νομίζω ότι έτσι προγάγονται οι διαπραγματεύσει. Μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν τέτοιε δηλώσει. Και νομίζω ότι αυτά κατατρέφουν και το κλίμα εμπιστοσύνη. Και το δηλώνω αυτό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να καταρτήσουμε νομοθεσία κανονισμό που να είναι αντίθετος στα συμφέροντα του κλάδου. Θα το προσπαθήσουμε. Εγώ δεν ε, λέω ότι δεν υπάρχει ελπίδα να πετύχουμε κάτι στα πλαίσια της Μαλτέζικης Προεδρίας, μόνο όμως αν υπάρχει και κάποια πρόοδος, μια κίνηση προς ε, τη μεριά μας. Ιντάλλως σας περιμένουμε τι έχει να μας πει η Μαλτέζικη Προεδρία. Αυτό είναι το πνεύμα των τριμερών διαλόγων. Άλλωστε, το να γίνουν συμβιβασμοί. Και το δηλώνω ευθερασώ ότι από την άλλη πλευρά δεν έχουν γίνει επαρκεί συμβιβασμοί. Ευχαριστώ, Ρε Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στον γύρο των ερωταπαντήσεων. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τους 14 τριμερείς διαλόγους που έχουν ήδη γίνει, να σας πω ότι εγώ συμμετείχα και πραγματικά επιβεβαιώνω κάποια από τα πράγματα που είπε ο κύριος Χόισλινγκ, ο συνάδελφος. Νομίζω ότι όλοι και αυτό το καταδεικνύει και η χθεσινή εκδήλωση. Όλοι μας λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα καταφέρουμε στην τελική ανάλυση. Ιδανικά, υπό τη Μαλτέζικη Προεδρία να πατήχουμε ένα συμβιβασμό, μια συμβαστική συμφωνία. Δεν είναι και πολλά ανοιχτά τα, δεν είναι και πολλά τα ανοιχτά και κρεμή στοιχεία έχουν καταφέρει να λύσουν πολλά θέματα οι προηγούμενοι τρέμερες διάλογοι. Και νομίζω ότι επί της ουσίας πλέον δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και χάρη σε αυτή την έλλειψη πολιτική βούληση δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν έχει και νόημα τώρα να μην κάνουμε τίποτα μέχρι τις 22 Μαρτίου, οπότε προγραμματίζεται και η επόμενη ε, συνάντηση στα πλαίσια τρομερού διαλόγου. Και μετά τον Απρίλιο και τον Μάιο να κάνουμε άλλο έναν τρίμερη διάλογο και τελικά να καταλήξουμε στην ίδια ακριβώς, ε, λίγο πολύ μάλλον, ε, κατάσταση το Σεπτέμβριο. Άρα, Μέχρι τις 22 Τρίτου θεωρώ ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές βήμα για συμβιβαστική διάθεση. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να αφήσουμε κατά μέρο την προσπάθεια αυτή τώρα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα αύριο κατά την παρουσίαση του Πρόεδρου Μάρτη να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες παρουσιάσεις και απολογισμούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμμετείχα, είχα την τιμή να συμμετάσχω σε αυτούς τους 14 τριμερείς και ευχαριστώ τον κύριο Χόισλινγκ γιατί είχε μεγάλη υπομονή και ήθελε πραγματικά να φτάσουμε σε συμβασμούς. Νομίζω ότι είδαμε και τα ετούμενα του τομέα και νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία για να φτάσουμε σε αίσιο πέρας ως προς αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να γίνει μία έρευνα για να τα καταφέρουμε στην έκθεση αυτή αξιοπρεπώς. Νομίζω ότι δείξαμε τη συνέπειά μας ως Κοινοβούλιο του τριμερείς και θα πρέπει η Προεδρία της Μάλτας να κάνει μία προπαρασκευαστική εργασία και να φτάσει στους ε, τριμερείς με μια πραγματική εντολή διαπραγματεύσεων που να συμμερίζεται η πλειοψηφία των κρατών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τέλος, δεν θέλω να μακρηγορήσω, υπήρχαν και σημεία σκληρής διαπραγμάτευσης ως προς τους ελέγχους και τα ε, κατόφλια που, όπου βρισκόμαστε πολύ κοντά με τον ε, από κοινού ε, νομοθέτη, με τον συνομοθέτη. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας ε, συνοδεύσει σε αυτή την πορεία και να μην έχουμε δύο συνομοθέτες που δεν εναρμονίζονται. Θα πρέπει λοιπόν σε μια διαδικασία παύσης να ορίσουμε το ρόλο του καθενός για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Γιατί τώρα ο τομέας περιμένει μία διέξοδο. Είναι ένας τομέας που περιμένει νέους κανόνες σε σχέση με τη βιολογική δηλαδή παραγωγή και γι' αυτό νομίζω ότι και οι τρει υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι, θα πρέπει να ορίσουν μία κοινή μέθοδο εργασίας. Gerling. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ παρευρέθηκα στους 14 τριμερείς από το ECR και είχαμε αυτές τις συνήθεις ενημερώσεις λίγο βαρετές θα μπορούσα να πω και ίσως η τακτική μας δεν είναι και τόσο δυναμική. Φτάνουμε στην αναπόφευκτη θέση ε, που συμβαίνει συχνά όταν πρόκειται για ένα τέτοιο νομοθετικό θέμα όπου γραμμή προς γραμμή θα πρέπει κανείς να δει όλα αυτά τα βιολογικά προϊόντα ένα προς Θα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε στα τελικά στάδια της διαπραγμάτευσης και στο τέλος των τριμερών υπήρχε η τάση συνένεσης από τα τρία θεσμικά όργανα δεν πρέπει να πούμε ότι εμείς κάναμε συμβιβασμό ενώ το Συμβούλιο δεν το έκανε. Εμείς αργήσαμε, καθυστερήσαμε νομίζω και με βάση το χρονοδιάγραμμά τους το γεγονός θα πρέπει να γίνει αναπομπή στις συνεδριάσεις τους και να ξαναέρθουν δεν μπορούσαν να παραδώσουν έργο και το ξέραμε αυτό τα ξέραμε αυτά εξ αρχής, άρα θα πρέπει να μην είμαστε αυτάρεσκοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εργασία κάθε αυτή. Συμφωνώ με τον κύριο Λίντς ότι θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά στο παρασκήνιο για να φτάσουμε σε αυτά συμπεράσματα και αποτελέσματα στον επόμενο τριμερή διάλογο και να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στον εισήγητη. Μας είπε ότι συναντήθηκε κατηδία με τους Μαλτέζους, αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης ο Σκιώδης. Ξέρω ότι στο τέλος του τελευταίου τριμερούς έκανα ορισμένες υποδείξεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά δεν έλαβα απαντήσεις. Εάν λοιπόν θέλουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, να κινηθούμε επαγγελματικά, εγώ θα συνενέσω. Και αυτό αφορά και τη συνάντηση με τον τομέα αυτό, με τον τομέα όπου δεν είχαμε δυστυχώς μια μεγάλη προθεσμία. Το μάθαμε τελευταία στιγμή. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο την Αυστρία και τη Γερμανία. Είναι ένας κανονισμός που αφορά τους πάντες. Και θα πρέπει να καλείτε τους ανθρώπους, να τους δίνετε χρόνο, να μπορέσουν να παρευρεθούν στις Βρυξέλλες. Δεν μπορείτε να μας το λέτε την προηγούμενη μέρα ή δύο μέρες πριν για να πρέπει να έρθουμε στις Βρυξέλλες για τις συναντήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταντέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση καθώς και τον σκιώδη της ομάδας μας που κατέβαλε πολύ μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Όπως ε, εδώ και 18 μήνες ε, Ίσως και λίγο περισσότερο εγκρίναμε αυτό το κείμενο, είχαμε πολλά μπρος πίσω πολλές παλινοδίες και δεν ξέρω κατά πόσο η συγητής θα μπορούσε να ζητήσει, να γίνει μια συνάντηση με όλους τους βοηθούς μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα υπόμνημα για να ανοιχνεύσουμε όλα τα σημεία, γιατί ε, δυστυχώς το κείμενο είναι σχηνοτενές, κάτι το οποίο δημιουργεί απορίες στον τύπο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δηλητηριάσουμε περισσότερο την ατμόσφαιρα από ό,τι ήδη είναι. Ο κ. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Και από πλευρά μου θα ήθελα να πω να ευχαριστήσω τον σκιώδη και τους σκιώ, τον, τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Θέλω να επανέλθω όμως ένα θέμα, γιατί έχω λίγο το δυσάρεστο συνέστημα ελπίζω να κάνω λάθος, ότι τώρα θα καταλήξουμε σε ένα ψεύτικο συμβιβασμό. Και αυτό θα σήμερα ότι όλα θα μείνουν όπως έχουν σήμερα. Ότι τα τρόφιμα δηλαδή, που παράγεται στην Ιταλία, ένα τρόφιμο που παράγεται στην Ιταλία, το οποίο χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα στα όρια, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ένα γερμανικό αυστριακό προϊόν μπορεί να, να κυκλοφορήσει και να τη χάνει εμπορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και αυτό δεν έχει να κάνει με την ενιαία αγορά καθόλου. Έχουν επιμείνει πολύ έντονα οι χώρες στις θέσεις τους Ακούσαμε τον Γερμανό Υπουργό Γεωργίας και να σας πω ότι και ο δικός μου υπουργό από την Ιταλία τα ίδια ακριβώ λέει, μόνο αντίθετα. Νομίζω ότι η χειρότερη δυνατή λύση θα ήταν να συνεχίσει να υπάρχει μια κατάσταση όπου υπάρχουν για τα ίδια προϊόντα άλλες προδιαγραφές παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και όπου, για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή αγορά θα είναι άδικη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην καταλήξουμε σε μια τέτοια συμβαστική λύση. Να κάτσουμε να σκεφτούμε αν ένα προϊόν βιολογικής παραγωγής θα πρέπει να έχει πραγματικά τις ίδιες τιμές όπως ένα συμβιωτικό προϊόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ειλικρινείς. Και σε κάθε περίπτωση ο σωστός συμβασμός θα είναι κάπου στη μέση, μια χρυσή τομή. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια ενδιάμεση, μια κοινή λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωστίνγκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσοντα και να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Πολλά ακούσαμε ήδη και εγώ πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά και ωριακέ μέση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα τον ε, οικονομικό κλάδο, το γεωργικό κλάδο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την πολιτική άποψη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Και η κυρία Γκέρλινγκ πολύ σωστά είπε το εξή. Δεν είναι μόνο για τη Γερμανία και την Αυστρία ο κανονισμό. Είναι σημαντικό να κοιτάξουμε πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση σε όλα τα κρατημέλη, για να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Και θα ήθελα να θίξω το θέμα και των εισαγωγών. Εν μέρει φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις ε, εξακολουθούν να θέλουν ιδιαίτερους τις φθηνές ε, εισαγωγές. Εγώ νομίζω όμως ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα βλάψει ιδιαίτερος τον ε, κλάδο βιολογική παραγωγή, γιατί θα χάσει την αξιοπιστία του και θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν διαρκώ να προσπαθούμε να εξισώσουμε προ τα κάτω το επίπεδο. Το θέμα που θέλω να θίξω επίση είναι το θέμα των σπόρων. Και εδώ πρέπει να σα πω ότι ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Ο κλάδο αυτό πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι ελκυστικό να χρησιμοποιεί κανείς βιολογικούς σπόρους αν δεν δώσουμε κίνητρα, δεν θα συμβεί τίποτα στο μέλλον. Και αυτή η δικαιολογία ότι αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν στον κανονισμό για τους πόρους μας κάνουν να γελάμε. Θυμάμαι το 2013 όταν μας υπέβαλαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπής ένας κανονισμός ε, για τους σπόρους ε, και τότε ένας κλάδος αντιτάχθηκε σύσσωμος. Άρα, αν το αποφύγουμε πάλι, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Μάκρο πρόθεσμα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε οι βιολογικοί σπόροι να είναι βιώσιμοι και να αξίζουν τον κόπο. Να έχουν ένα κίνητρο για αυτά που είπε ο κ. Χόισλινγκ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι στην κριτική Τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά, άλλωστε, στη Γεωργία. Δεν πρέπει να αντιδρούμε με προβολικό τρόπο. Το οφείλουμε αυτό και στους ε, καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, γιατί ήδη καταβάλουν μία προσπάθεια και θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει το κλάδος αυτός. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Γιάρ. Καταρχάς, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους και Δεν ήταν εύκολο το έργο που είχα να κάνω. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση έχω να κάνω. Έχω σχεδόν την εντύπωση ότι δεν θέλει συμφωνία το Συμβούλιο. Δεν το ενδιαφέρει. Ότι η διάθεση που επικρατεί είναι ότι από το να πετύχουμε κάτι κακό, ας ε, μην πετύχουμε τίποτα ο κ. Χόισλινγκ μα είπε με καλή παρουσίαση το τι παραμένει κρεμές και ανοιχτό. Οι ωραίε τιμέ Θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως σημείο κίνησης και για τα υπόλοιπα προβλήματα. Να υπάρξει κάποια κίνηση, εν περιπτώσει. Μήπως είναι αυτό το κλειδί. Αυτό θα ήθελα να απευθύνω σε ερώτηση στον κύριο Χόισλινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε να Δεν να λάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, γιατί με τα πιο πολλά συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι επί τη αρχή πρέπει να πούμε το εξή. Αν μια διαδικασία ψήφιση μια οδηγία, έχει πάρει 12, 18 μήνε, και δεν υπάρχει και οποιαδήποτε τέτοια προοπτική στην παρούσα φάση, αυτό ήδη βλάπτει πάρα πολύ τον κλάδο. Αυτό πραγματικά είναι πολύ αρνητικό και θεωρώ ότι οφείλεται στην αδυναμία και την απροθυμία μάλλον του Συμβουλίου να κάνει συμβιβασμό. Και στο θέμα των συμβιβασμών από το εξή. Αν τελικά ο συμβιβασμό είναι κακός, θα πρέπει να έχουμε την ε, τόλμη να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις και Αγαπητέ κύριε Χόισλινγκ, έχετε λάβει από εμάς μια σαφή εντολή. Και στο πλαίσιο τη εντολής θα πρέπει να κάνεις τι διαπραγματεύσει. Αν δεν είναι αυτό δυνατόν, θα πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται αυτό που πλευρά στο Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σαγνιό. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καιρό μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς τον Μάρτιν Χάουσλινγκ. Γιατί με πίεσαν πάρα πολλοί οι Σκανδιναβοί γεωργοί, οι οποίοι ανησυχούν για το γεγονός ότι τελικά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνανε, δηλαδή να καλλιεργούν σοδιές ε, σε πάνω από τη γη, ας πούμε, ε, που να μην παγώνουν κτλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Ε, μιλάμε για την συνέχεια για την καθαρότητα των βιολογικών καλλιεργικών που δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου φυτοφάρμακα. Εγώ σημείωσα. Ε, επιτρέπεται σε 30 τόνους ε, ε, ε προϊόντων να έχουμε ε, διάφορα πράγματα, ε, ας πούμε ρινίσματα ξύλου, ε, έντομα, ε, διάφορα πράγματα μέσα. Δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη καθαρότητα στη γεωργία. Επίσης, κανένας δεν με πίεσε, δεν με πίεσαν οι Βρετανοί ε, καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων τα τελευταία δύο χρόνια δεν με ενόχλησαν καθόλου. Επομένως, διερωτώ με, τελικά τι χρειαζόμαστε αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το σημείο, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για αυτό το έγγραφο. Τώρα ακούμε διάφορα πράγματα. Επομένως, κύριε Νόχελ, εάν έχετε χρόνο σε επόμενες συζητήσεις, να λάβετε υπόψη σας ότι ο κλάδος δεν έχει καμία ασφάλεια για την κατάστασή του. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το σημείο αυτό στην Προεδρία και ίσως ε, οι συγητές θα μπορούσαν να βάλουν αυτό το θέμα σε ένα γραπτό κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να φτάσει στους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Κυρία Κιώστιγκερ. Για το θέμα αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια. Νομίζω ότι κατά 90% του κανονισμού την έχουμε διαπραγματευτεί. Όλα. Ε, είμαστε, έχουμε κάποια σημεία που μας προβληματίζουν ακόμα. Τώρα, να τα πετάξουμε όλα στα σκουπίτια για το 10% που έχει απομείνει είναι κρίμα. Και δεν θέλουμε να επανέλθουμε στο status quo. Και ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες, διάφορες οργανώσεις που θα το καλωσόρισαν αυτό το να παραμείνει το status quo. Αλλά δεν θα ωφελούσαμε τους γεωργούς και τους εκτροφείς. Το οφείλουμε λοιπόν και στους γεωργούς και στους καταναλωτές να αναπτύξουμε αυτό το μέσο και να το κρατήσουμε λειτουργικό για να μπορέσει να έχει νόημα η βιολογική καλλιεργία για στο μέλλον. Μάλιστα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι δεν θα ασχοληθώ με το θέμα Θεωρώ ότι με καλή θέληση μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις κάπου. Κύριε Χόισλιν. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο ενδελεχώς αυτά με τις ομάδες, αλλά συμφωνώ με την κυρία Κώστινγκερ ότι ως τώρα έχουμε κάνει τη δουλειά κατά 80%. Θα ήταν καλό να γίνουν αποδεκτές ε, οι συμβασικές προτάσεις από το Συμβούλιο και αναφέρθηκαν διάφορα θέματα. Το θέμα των ε, φυτοφαρμάκων όπως το έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, βρίσκει σύμφωνο ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο. Αυτό είναι σαφές ως, είναι σαφές ως θέση. Και άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν το σύστημα ελέγχου των κοινωνικών προτύπων. Στόχος θα πρέπει να είναι στον κανονισμό αυτό να υπάρξει καταρχά μια ευρωπαϊκή ενερμόνιση. Αυτή είναι η ουσία. Δεν μπορούμε να έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα και να εφαρμοστούν αυτά με διαφορετικό τρόπο. Και εδώ συμφώνω με την κυρία Κέρστιγκερ. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει πιο ακριβό, πιο ακριβή η βιολογική σπόρη. Ενισχύουμε λοιπόν τα μέτρα πρόληψη και εδώ θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και ο οικονομικό κλάδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να μα υποβάλει μια έκθεση για το status quo και το 2020 και τώρα θα έχουμε και τότε θα έχουμε κάτι στα χέρια μα. Το χειρότερο θα ήταν να μείνουν τα πράγματα και να παγώσουν όπως έχουν τώρα. Γιατί ξέρετε το χρονικό περιθώριο περιορίζεται και πάει. Εγώ δεν θέλω μία διαπραγμάτευση χωρίς τέλος. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τρεις, άντε τέσσερις τρεμερείς διαλόγους στην Μαλτέζικη Προεδρία και μετά να πούμε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία, δυστυχώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία. Ενδεχομένω όμω και στα άλλα κρίσιμα σημεία να μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία. Συμφωνώ αυτό που είπατε μόλι για το θέμα των ε, εισαγωγών. Να μην υπονομεύσουμε τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα και να αποδεχτούμε πρότυπα τα οποία είναι χαμηλότερα από αυτά που συζητάμε από τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα να επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε όλο τον κλάδο και αυτό θα πρέπει να το συνηθίσει και να το εφαρμόσει και ο οικονομικό κλάδο. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο ότι κάτι καταφέρουμε. Αλλά το να καταλήξουμε σε έναν οποιοδήποτε συμβιβασμό, μόνο και μόνο για να υπάρχει συμβιβασμό, δεν πρόκειται να με βρει σύμφωνο. Καλύτερα να μην έχουμε καθόλου συμβιβασμό. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τα κρατημέλη. Γι' αυτό λοιπόν ας συνεχίσουμε τη δουλειά μας και όπως σας είπα, δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε μέχρι το τέλη Μαρτίου. Ως Κοινοβούλιο θα παρουσιάσουμε την διαπραγματευτική μας θέση προκειμένου να καταφέρουμε να περάσουμε στο τελευταίο ετάπ την από τέλη Μαρτίου. Να συνεχίσουμε και τις συζητήσεις ε, με τον γεωργικό κλάδο και να σας πω ότι χθες οι συζητήσεις μας με τον οικονομικό κλάδο επιβεβαίωσαν πολλάκις τη θέση μας. Και θεωρώ ότι αυτή την ορμή θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και στις διαπραγματεύσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Χόισλικ, να σας ρωτήσω το εξής. Όταν θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, ίσως θα γίνει λόγος για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Πώς μπορούμε ας πούμε, να προσεγγίσουμε τα πολιτικά κόμματα για να πετύχουμε τη συμφωνία. Και κυρίως πριν τις 23 Μαρτίου τι πρέπει να γίνει τόσο ώστε να συζητήσουμε ξανά το θέμα στην Επιτροπή μας. καλό θα ήταν μετά από αυτές τις θέσεις που ακούσατε από τα μέλη της Επιτροπής μας να διαμορφώσετε τη θέση σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταματάμε τώρα εδώ. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στη συνεδρίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 6.30 έχουμε μια συνεδρίαση με τους νέους γεωργούς. Και τώρα θα κάνουμε δύο λεφτά τεχνικό διάλειμμα και σε δύο λεφτά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών.